Και φτάνω στην ημερήσια διάταξη των εργασιών μας. Με βάση την απόφαση της σκέψης των Προέδρων δυνάμει του άρθρο 159 του κανονισμού έχει διανεμηθεί και σε συνεργασία και συμφωνία με τις ομάδες προτείνω καταρχάς... Όχι, σας είδα. Σε συνεργασία με τις ομάδες προτείνω η ψηφοφορία για τις εκθέσεις της κοινή συζήτηση για την κοινή πολιτική ασφάλειας και, άμυνα, και άμυνας να αναβληθούν για την πέμπτη την ώρα των ψηφοφοριών δηλαδή για δε την κατεξοδότηση πρόταση κανονισμού για τον κανονισμό ε, γεωργικής προέλευσης από την, αντί για την πέμπτη να έρθει πιο νωρίς την τετάρτη η ψηφοφορία. Τετάρτη λοιπόν τα γεωργικής προελεύσεως αλκοολούχα. Βλέπω ότι συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών υποστήριζε την αλλαγή αυτή. Η κυρία Τσούπε έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Απλώς να σας πω ότι την προηγούμενη Παρασκευή ο πρόεδρος Ποροσέγκο ε, ενέκρινε μία σειρά νομοθετημάτων που αποτρέπει και καταργεί τη χρήση των ε, σημάτων του κομμουνιστικού καθεστώτος και ήθελα να μου πείτε τι προτίθεστε να κάνετε. Ευχαριστώ, πλέον όμως αυτό δεν έχει σχέση με την ημερήσια διαταξή μας. Ο κύριος Βιώτη νομίζω έχει στο στολό. Παρακαλώ. Σήμερα το πρωί ο Ιταλικός τύπος αναφέρεται στο εξής. Στη Βουδαπέστη υπάρχει ένας νέος 33 ετών που ε, μπορεί να, να σκοτωθεί γιατί είναι ακτιβιστής γκέι και η πληροφορία αναφέρθηκε από το κόμμα Γιόμπικ. Έχει επικηρυχθεί με 10.000 και είναι απαράδεκτο μια ευρωπαϊκή χώρα να απειλεί ένα νέο παιδί επειδή είναι ακτιβιστής γκέι. Την επόμενη, τον επόμενο Ιούλιο θα γίνει η παρέλαση Pride και θα ήθελα όλοι να βρεθούμε στο, στη Βουδαπέστη για να καταδικάσουμε αυτή την τάση. Ωστόσο, δεν έχει σχέση αυτό με την ημερησία μας διάταξη τη σημερινή, κύριε Ποιώτη. Και Δευτέρα. Σήμερα υπάρχουν παρατηρήσεις για την ημερησία διάταξη. Όχι. Τρίτη, η ομάδα των Πρασινών και των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ζητούν Συζήτηση για Η συζήτηση για την κατάσταση στην Ουγγαρία με δηλώσει του Συμβουλίου και τη Επιτροπή να ολοκληρωθεί με ψήφισμα. Η δε ομάδα των Πρασίνων ζητεί και ονομαστική ψηφοφορία εν προκειμένου. Δίνω το λόγο στην κυρία Χάρμς. Πρόεδρε, η ομάδα μου Ήδη από την προηγούμενη ε, και τις δηλώσεις του Βίκτορ Όρμπαν για την θανατική ποινή στην Ουγγαρία έχει ζητήσει να συζητηθεί σοβαρά το θέμα αυτό. Υπάρχει ένα ζήτημα ε, πρότασης από την κυβέρνηση για διευκρίνηση του θέματος, η λύση του θέματος των μεταναστών με δημοψήφισμα. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να αντιδράσουμε. Ήδη από την έκθεση Τάβαρες έχουμε επισημάνει ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην Ουγγαρία. Ο Βίκτορ Ουρμπάν ε, καταχράται τις πλειοψηφίες που έχει στη χώρα προκειμένου να παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα και αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι πρέπει να αντιδράσουμε αυτό και την ερωτική αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη χρειαζόμαστε όχι μόνο για το Fiscal Compact, για τα δημοσιονομικά μέτρα, αλλά και για να αντιδρούμε σε θέματα ανθρωπινών δικαιωμάτων και αξιών. Πρέπει να τα συστήσουμε λοιπόν και να τα καταγράψουμε σε ένα ψήφισμα. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ εκ των και Δημοκρατών, ο κύριος Κερίρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω περισσότερο για το κατά πόσο χρειάζεται ή δεν χρειάζεται ψήφισμα, γιατί συμφωνώ με τα όσα είπε η κυρία Ρεμπέκα Χάρμς πριν από λίγο. Το θέμα είναι ότι η ομάδα μου θα επιθυμούσε το ψήφισμα αυτό να οριμάσει μετά τη συζήτηση που θα έχουμε αύριο το απόγευμα. Και συνεπώς προτιμούμε το ψήφισμα να ψηφιστεί τον Ιούνιο. Ναι, ψήφισμα, αλλά κατά προτίμηση τον Ιούνιο. Πριν εκθέσω στη συζήτηση και ψηφοφορία τις προτάσεις αυτές, θέλω να επισημάνω τα εξής διαδικαστικά. Η Λετωνική Προεδρία με ενημερώνει με επιστολή από 14 Μαΐου ότι δεν σκοπεύει να λάβει μέρος στη συζήτηση αυτή γιατί δεν υπάρχει ενιαία τοποθέτηση του Συμβουλίου. Ταυτόχρονα, ο, πρόεδρος, ο Πρωθυπουργός Ορμπάν μου αποστέλει επιστολή ο οποίος με παρακαλεί να με την οποία με παρακαλεί να επιτρέψω τη συμμετοχή του στη συζήτηση εδώ. Διαδικαστικά θα ενημερώσω αποκλειστικά διαδικαστικά και μόνο θα ενημερώσω ότι δεν γνωρίζω να υπάρχει προηγούμενο που η Προεδρία να απορρίψει ή να αρνηθεί τη συμμετοχή της σε συζήτηση με επιχείρημα ότι δεν υπάρχει κοινή θέση του Συμβουλίου για το θέμα. Μια σειρά από νομοθετήματα συζητήθηκαν ε, και λέγαμε «Α, θα πρέπει να έχει πάει διακοπές στο Συμβούλιο». Δεν μπορεί να είναι αυτό επιχείρημα. Ο Πρωθυπουργός Ορμπάν ασφαλώς και θα προσκληθεί από τον πρόεδρό σας, εφόσον το επιθυμείτε να έρθει εδώ. Ο κανόνας που τηρούμε πάντα είναι ότι μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου βεβαίως και αυτονόητα μπορούν να επισκέπτονται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να υποστηρίζουν τις θέσεις τους εφόσον το επιθυμούν. Το έχουμε καταστήσει σαφές αυτό και εν ώψη της ευρωπαϊκής πολιτικής, το έχουμε επανελειμμένως δηλώσει, εφόσον το επιθυμεί ο κ. Σουρβάν. Αλλά, αλλά δεν επιτρέπεται να έρθει ο κύριος Ορμπάν για να διαδραματίσει το ρόλο της Προεδρίας εδώ. Στο βαθμό αυτό λοιπόν πρέπει να ορίσουμε διαδικαστικά τον τρόπο εργασίας μας και γι' αυτό καλώ τους προέδρους των ομάδων να έρθουν ε, μέσω με τα την εργασιών, ε, με το που θα αποχωρήσω, στο γραφείο μου για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε διαδικαστικά την αυριανή παρουσία του κύριου Ορμπάν. Ε, για την ουσία τώρα, ακούσατε την κυρία Χάρμς, ακούσατε τον κύριο Γκερέρο. Ε, ποιος είναι υπέρ των προτάσεων. Ποιος είναι υπέρ της πρότασης Πρασίνων και Σουριστών Δημοκρατών. Κύριε Νετφέλτ. Ευχαριστώ. Η ομάδα μου στηρίζει την πρόταση των Πρασίνων. Στηρίζουμε επίσης το ψήφισμα να γίνει το Μάιο, γιατί το είπατε κι εσείς. Υπογραμμίζει το πόσο επίγον είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφανθεί επί του ζητήματος αυτού. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν πρέπει να καθυστερήσουμε. Οπότε στηρίζω την πρόταση. Καλώς λοιπόν. Έχουμε να κάνουμε δύο Κυρία Χάρμς, περιμένετε ένα λεπτό παρακαλώ. Έχουμε να κάνουμε δύο ταυτόσιμα αιτήματα, ε, δηλαδή συζήτηση με ψήφισμα, αλλά διαφορετική διάσταση προς το χρόνο, γιατί οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες ζητούν να γίνει τον Ιούνιο, τώρα εσείς όμως επιμένετε για τον Μάιο. Μάλιστα, ποιος είναι κατά της προτάσεως, ο κύριος Ζάιερ. Νομίζω ότι Νομίζω ότι η διαδικασία που γίνεται τώρα κάποιον που δεν ανήκει στην πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λέει κάτι και λέμε κατεπηγόντως συζήτηση και ψήφισμα δεν είναι καλό. Η Ρεβέκα Χάραμς έδωσε δύο επιχειρήματα γιατί πρέπει να έχουμε ψήφισμα και τα δύο είναι εσφαλμένα. Το πρώτο, για παράδειγμα, ο ίδιος ο κύριος Ορμπάν στη συζήτηση που είχε με την Προεδρία αλλά και δημόσια είπε ότι δεν παίρνει μέτρα για να επανεισαγάγει τη θανατική ποινή. Το άλλο θέμα είναι το κατά πόσο θα υπάρχει δημοψήφισμα ή στην Ουγγαρία. Μα δεν υπάρχει δημοψήφισμα στην Ουγγαρία. Η κυρία Χάρμ ζητάει ψήφισμα γι' αυτό, θα έπρεπε όμω να έχει προετοιμαστεί καλύτερα. Γιατί δεν πρόκειται για δημοψήφισμα, πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο για το θέμα της μετανάστευσης, που είναι το καυτό ζήτημα στην Ευρώπη σήμερα. Δεν θέλουν να ερωτηθούν οι άνθρωποι για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, τα δύο επιχειρήματα της κυρίας Χάρμς είναι εσφαλμένα, γι' αυτό και εγώ λέω να μην έχουμε ψήφισμα για αυτό το θέμα. Ich muss Θα πρέπει να επιβεβαιώσω το ορθό κομμάτι της τοποθετήσεως από αυτή τη θέση. Με προλάβατε κύριε Ζάιερ, γιατί είχα δηλώσει από την προηγούμενη σύνοδο ότι θα τηλεφωνούσα με τον στον κύριο Ορμπάν, μιλήσαμε για πολλή ώρα, μου εξήγησε ακριβώς αυτό το οποίο μας εξηγήσατε εσείς κύριε Ζάιερ, ότι δεν έχει διάθεση, δηλαδή η πρόθεση η κυβέρνηση να λάβει ε, διαδικασία δημοψηφίσματος και να εισαγάγει θανατική ποινή. Αυτό άλλωστε το δημοσίευσαμε και σε ένα ανακοινωθέν τύπου. Για να είναι ε, τώρα λοιπόν, ψήφισμα νέου ψηφίζουμε και για τη χρονική στιγμή. Πρώτα όμως ψηφίζουμε για το ποιος θέλει ψήφισμα μετά δημοψηφίσματος. Είπε κατά. Πλειονοψηφία νομίζω. Ας επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Τώρα ψήφισαν όλοι. Πέρα τις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Τώρα, το ψήφισμα για το Μάιο, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Ε, ήταν σαφέ πως πρόκειται για πλειοψηφία. Τώρα, τον Ιούνιο το ψήφισμα. Ψήφισμα τον Ιούνιο υπέρ κατά. Ε, εγκρίνεται. Κατάθεση τροπολογιών. Θα οριστεί αναλόγως η προθεσμία δεδομένου ότι πρέπει να ψηφίσουμε τον Ιούνιο. Παρακαλώ. Πρόεδρε, θέλω να επιμείνω σε αυτό που είπατε για την παρουσία του Συμβουλίου. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά το ξέρετε ότι πολλές φορές στην Επιτροπή Ελευθερίων του Πολίτη η Λετωνική Προεδρία έχει την ίδια στάση. Νομίζω λοιπόν ότι είναι συνολικό το πρόβλημα. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με ορθό τρόπο. Το Συμβούλιο δεν σέβεται τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα εδώ και θέλω να επιμείνω πάνω σε αυτό παρακαλώ. Ich glaube, dass ich meine Position zu Νομίζω ότι κατέστασα σε αυτή τη θέση μου σε σχέση με την ε, συμπεριφορά του Συμβουλίου. Τετάρτη. Δεν έχω προτάσεις για τροποποίηση. Πέμπτη. Η ομάδα σοσιαλιστών και δημοκρατών προτείνει να γίνει το πρωί η συζήτηση για τα θέματα των ανθρωπινών δικαιωμάτων και να γίνει ψηφοφορία στις 12. Ο κύριος Γκερέρο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ομάδα μου, γενικά μιλώντας, θα ήθελε οι συζητήσεις για τα κατεπήγοντα να γίνονται πάντα την Πέμπτη το πρωί. Και αυτό για να τους δώσουμε την σημασία που πραγματικά έχουν τα θέματα αυτά που συζητάμε στα κατεπήγοντα. Μερικές φορές τελικά κανένας δεν ενημερώνεται. Είναι μια γενική θέση. Οπότε αυτό που ζητάω είναι αυτή την ολομέλεια, τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα κατεπήγοντα να συζητηθούν το πρωί και να ψηφιστούν στις 12 το μεσημέρι. Υπέρ της προτάσεως, ποιος θέλει να λάβει το λόγο, κάνεις. Κατά, κύριε Πρέντα. Δεν συμφωνώ με την ιδέα του να συζητηθούν τα κατεπήγοντα το πρωί για δύο λόγους. Καταρχήν, γιατί την Πέμπτη το απόγευμα μπορούμε να εργαστούμε άρτια. Δεν βλέπω γιατί πρέπει να εργαζόμαστε τρεις ημέρες και όχι τέσσερις πλήρεις ημέρες και ήδη υπάρχει η παράδοση του Κοινοβουλίου να ασχολούμαστε με τα κατεπήγοντα το απόγευμα και συνήθως ο κόσμος είναι πολύ περισσότερος από όταν προγραμματίζονται για το πρωί της Πέμπτης. Άρα αντιτίθεμε στην πρόταση των σοσιαλιστών. Okay. Καλώς. Κυρίε και κύριοι, ψηφίζουμε την πρόταση του κυρίου Γκερέιρο. Ποιο είναι υπέρ της προτάσεως του κυρίου Γκερέιρο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 185 υπέρ, 106 κατά. Εγκρίνεται η πρόταση. Okay.